Well, good Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω τα μέλη και το ακροατήριο στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Φορολογικά μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή δεν αδρανούσε, μια αντιπροσωπεία μας πήγε σε αποστολή στη Ουάσιγκτον τον Ιούλιο. Και άλλη αντιπροσωπεία πιο πρόσφατα πήγε στην ε, Λετωνία. Και έτσι πήραμε πρώτο χέρι πληροφορίες και στοιχεία για πολλά από τα στοιχεία που μας αφορούν. Θα συζητήσουμε ψηφιακή φορολόγηση σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι η αδελφή μας Επιτροπή, η ΕΚΟΝ ασχολείται με δύο νομοθετήματα. Στόχος τους η εξασφάλιση ότι οι ψηφιακές εταιρείες δεν ξεφεύγουν όσον αφορά τη φορολόγηση. Στην αποστολή μας στην Washington, D.C., η ψηφιακή φορολόγηση ήταν από τα θέματα που ενδιέφερε τους ομολόγους μας. Ήταν πολύ ζωρές συζητήσεις. Η ακρόαση θα ωφεληθεί από τη γνώση που αποκόμισα να τις συζητήσει στα μέλη μας. Με τη σημερινή συζήτηση θα εφαρμόσουμε την εντολή μας συμβάλλοντας τις συζητήσεις περί φορολογήσεως της ψηφιακής οικονομίας. Είμαι ότι η σημερινή συζήτηση θα τροφοδοτήσει το έργο των νομοθετικών οίκων στο σχετικό τομέα. Η ακρόαση θα αποτελεστεί από δύο παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων. Ο ένας είναι από τον ΟΣΑ και δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έντουαρτ Φολσόντας από την Γενική Διεύθυνση Ταξούτ θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοδεύεται από τον κύριο Βάτ Βαν Ράιν από την DG ε, Taxud. Ο κύριος Έρικ Ρομπέ από τον ΟΣΑ θα παρουσιάσει τη θέση του φορέα για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Καλώς ήρθατε κύριοι στην συνεδρίαση. Θέλουμε να ακούσουμε τις παρουσιάσεις σας. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας σχετικά με την ψηφιακή φορολόγηση. Κάθε θεσμικό όργανο θα έχει ένα δεκάλεπτο για παρουσίαση. Μετά την παρουσίαση από τους ομιλητές θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων. Κύριε Φολσόγκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Μπάρτ και εγώ είμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετοιμάζουμε το πακέτο για την ψηφιακή φορολόγηση. Δοθέντων των χρονικών περιορισμών, θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε κάποια σημεία, τις βασικές πτυχές του πακέτου. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που συζητούνται. Αν κάποια από τα θέματα δεν καλυφθεί στην παρουσίασή μου, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε και να το τονίσετε σε ερωτήσει. Θα καλύψω ακροθυγό το πρόβλημα προ επίλυση. Μετά ακροθυγό θα περιγράψουμε τις λύσεις που διαφαίνονται και που προτείνουμε. Να τονίσω κάτι. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Επιλύεται από διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι θέλουμε να λύσουμε. Τη φορολόγηση εισοδήματο εταιριών και πώς εφαρμόζεται η φορολόγηση στο ψηφιακό τομέα. Έχουμε ψηφιοποίηση, που είναι ένα γεγονό και επιτρέπει σε όσοι βαθμίδες τη κοινωνίας να κινητοποιηθούν ψηφιακά. Αυτό είναι πολύ καλό. Ενθαρρύνουμε την ψηφιοποίηση. Και η ψηφιακή ενή αγορά είναι πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σαν πολίτες, σαν χρήστες, Όλοι δεχόμαστε ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει ωφέλη. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και τις εταιρείες και τους κανόνες για φορολόγηση των εταιριών που έχουν θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια και περισσότερα για, τις, για τη φορολόγηση επιχειρήσεων και αυτοί οι κανόνες εδράζονται επί της ενίας της φυσικής παρουσίας. Δηλαδή μια εταιρεία πληρώνει άμεσα φόρους στη δικαιοδοσία, σε μια δικαιοδοσία αν είναι φυσικά παρούσα εταιρεία εκεί αν έχει έδρα εκεί, μόνιμη παρουσία εκεί. Διότι πριν από 100 χρόνια βλέπετε, αν μια εταιρεία ήθελε να κινηθεί σε μια αγορά, έπρεπε να είναι φυσικά παρούσα. Να έχει μια αποθήκη, να ανοίξει ένα κατάστημα. Γι' αυτό οι κανόνες βασίζονται πολύ επί της φυσικής παρουσίας. Αν συνδυάσουμε τις δύο πραγματικότητες, τι βλέπουμε, ότι δεν ταιριάζουν. Τα ψηφιακά επιχειρησιακά μοντέλα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά σε αόρατα, σε άειλα υλικά. Παράγουν την αξία, άειλη αξία. Και κλίμακα χωρίς μάζα, όπως λέει ο ΩΣΑ. Δηλαδή, από μακριά μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και να πλησιάζει τον καταναλωτή από μακριά. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις δεν έχουν έδρα για φορολόγηση σε μια δικαιοδοσία, συγκεκριμένη δικαιοδοσία, ενώ κινούνται επιχειρηματικά σε αυτή τη δικαιοδοσία και ωφελούνται από τις υποδομές ε, της ε, δικαιοδοσία χωρί να φορολογούνται από αυτή τη δικαιοδοσία. Γι' αυτό λέμε ότι το πλαίσιο τη φορολόγηση εταιριών είναι κάτι απερχιωμένο και οι ψηφιακέ επιχειρήσει δεν μπορούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματο εκεί που ε, επιχειρούν, λόγω των κανόνων που βασίζονται φυσική παρουσία. Όλε οι λύσει που προτείνουμε στο πακέτο ψηφιακής φορολόγησης προσπαθούν να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα από διαφορετική γωνία και σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Εδώ βλέπετε ότι τα προβλήματα που αναφέρουμε αναπτύσσονται, αυξάνονται. Γνωρίζετε το πολιτικό πλαίσιο, δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα αυτά. Συζητούνται εκτενώς. Εξετάστηκαν από τον ΩΣΑ, είχαμε πολιτική εντολή από το Συμβούλιο να τα επεξεργαστούμε και εμείς και να υποβάλουμε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου το Μάρτιο. Προτείνουμε λοιπόν αυτές τις λύσεις. Το πρόβλημα που περιέγραψα είναι παγκοσμίου εμβελίας και γι' αυτό χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η λύση. Τι εννοώ με αυτό. Μια λύση που θα συμφωνηθεί σε επίπεδο ΟΣΑ, σε διεθνές επίπεδο. Ε, ξέρουμε ότι αυτή η σφαιρική α, λύση χρειάζεται χρόνο για να είναι λογική. Είναι περιπλοκότατο το ζήτημα, βλέπετε. Η δομική λύση που πιστεύουμε που είναι η μόνη συνεπάγεται επαναπροσδιορισμό βασικών ενιών ε, μόνιμη εγκατάσταση κλπ. που φορά τη φορολόγηση των εταιριών. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τους κανόνες για την φορολόγηση των εταιριών σε επίπεδο της Ένωσης και προτείνουμε οδηγία για να αλλάξουν οι κανόνες που ισχύουν μεταξύ κρατών μελών και έχουμε και συστάσεις να αλλάξουν οι κανόνες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών Πρέπει να καθορίσουμε εκ νέου του κανόνε για τη φορολόγηση εταιριών, λαμβάνοντα υπόψη τον ψηφιακό παράγοντα. Δύσκολο το εγχείρημα. Χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό προτείνουμε βραχυπρόθεσμη λύση. Ε, προσωρινή λύση. Να εφαρμοστεί μέχρι την πλήρη λύση που θα εφαρμοστεί. Προσωρινό μέτρο. Ο, η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Η πλήρης λύση, θα την αναφέρω ακροθυγός αυτήν, έχει στόχο να αλλάξει την απάντηση σε δύο ερωτήσει. Αυτό που μας κάνει να Θα έχουμε δύο ερωτήσει. Όταν θέλουμε να καθορίσουμε τι φόρο πληρώνει μια, μια εταιρεία σε ένα κάτω μέλος. Τι φορολογούμε και πού το φορολογούμε. Για να πληρώσει άμεσους φόρους, εταιρικούς φόρους μια εταιρεία σε μια χώρα πρέπει να έχει φορολογική σχέση με αυτή την νομοθεσία. Αν βασίζεται η εταιρεία στη φυσική παρουσία, ε, δεν, υπά... αν δεν έχει φυσική παρουσία δεν υπάρχει αυτός ο φορολογικός δεσμός. Γι' αυτό προτείνω να δημιουργηθεί μια σχέση ψηφιακής φορολόγησης η εταιρεία για να, να πρέπει να καταβάλει φόρους σε ένα κάτω μέλο δεν είναι κάτι, δεν είναι απαραίτητο να έχει ψηφιακή, μόνο να έχει ψηφιακή μόνιμη παρουσία, αλλά θα πρέπει και τα κέρδη να μπορούν να σχετιστούν με αυτή τη μόνιμη ε, παρουσία, την ψηφιακή της εταιρεία σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό προτείνουμε να λάβουμε υπόψη την ψηφιακή πτυχή των επιχειρήσεων με τον τρόπο, στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει την κατανομή των κερδών. Αυτά βλέπετε. Τι προτείναμε. Πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Και από τη στιγμή που θα έχουμε καθορίσει ότι υπάρχει η ψηφιακή φυσική παρουσία θα πρέπει να γίνει κατανομή των κερδών σύμφωνα με τη λειτουργική ανάλυση που χρησιμοποιείται τώρα ενεργητικό κίνδυνος που αναλαμβάνει η εταιρεία και ψηφιακή πτυχή, κάτι που λείπει σήμερα. Πάω τώρα στο προσωρινό μέτρο. Αυτό που περιέγραψα, η πλήρης λύση, η τελική λύση, που πιστεύουμε ότι θα δώσει τα ακριβέστερα αποτελέσματα και θα είναι η ακριβέστερη λύση του προβλήματος, θα είναι μια ε, συμφωνία, θα χρειάζεται μια δύσκολη συμφωνία πρώτα. Εν τω μεταξύ έχουμε πιέσεις που ασκούνται πάνω μας να δράσουμε για προσωρινά μέτρα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης της φορολογικής ως στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποια αδικία που διαπιστώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε όσον αφορά τους κανόνες περιφορολογήσεως, διότι εντάσσονται στα παραδοσιακά κριτήρια αυτές οι εταιρείες και διαμαρτύρονται Συναντήσαμε αρκετέ ευρωπαϊκέ εταιρείε και μα είπαν ότι είναι σε μια θέση δύσκολη, δυσχερή, μειονεκτική επιχειρηματική, διότι αντιμετωπίζουν άλλε εταιρείε που δεν έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παίζουν με τι κανόνε. Έχουμε κατακαιρματισμό τη ενιαία αγορά, οπότε έχουμε και πρόβλημα συμμόρφωση. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να θεσπίζουν προσωρινά μέτρα. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί ότι οι προσωρινέ λύσει αποτελούν πραγματικότητα και χωρί δράση Ευρωπαϊκή Ενώση, ποιο είναι ο κίνδυνο. Ότι θα καταλήξουμε σε εμβαλωματικέ λύσει 28 προσωρινών μέτρων. Γι' αυτό προτείνουμε έμεσο φόρο, δυνάμει του άρθρου 113, όσον αφορά τα μεικτά κέρδη μέσω που προέρχονται μέσω ε, κάποιων ψηφιακών δραστηριοτήτων και μόνο. Μετά, γιατί προτείνουμε κάτι τέτοιο. Θα τεθεί και το θέμα του, της φορολόγησης κύκλου εργασιών αυτός απορρέει από τη φορολόγηση των κερδών και των εισοδημάτων των εταιριών. Γιατί προτείνουμε ένα φόρο κύκλου εργασιών. Αν θέλουμε προσωρινό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται τώρα, η αντιμετώπιση των κενών και διαφορών όσον αφορά τους κανόνες φορολογής εταιριών, αυτό το μέτρο το προσωρινό δεν μπορεί να συμμορφωθεί με του κανόνε που θέλουμε να αλλάξουμε. Και η φορολόγηση εισοδήματο θα έχει του ίδιου περιορισμού που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. μέσω μιας τελικής λύσεως. Τέλος, αυτό το προσωρινό μέτρο έχει, είναι πολύ στοχευμένο και από πλευράς των φορολογουμένων ατόμων, φυσικών προσώπων που πρέπει να καταβάλουν το φόρο και από πλευρά δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το νέο φόρο. Φορολογούμε μόνο κάποιες ψηφιακέ δραστηριότητες που βασίζονται πολύ στη συμμετοχή του χρήστη. Αυτή η συμμετοχή του χρήστη έχει νομισματική αξία, χρηματική αξία και είναι από τη βασική εισρωή για την παραγωγή κέρδους, εισοδήματο από τις Θέλουμε αυτό το δυναμικό να το αναγνωρίσουμε και γι' αυτό ο φόρος εφαρμόζεται σε αυτές τις δραστηριότητες με υψηλή ε, συμμετοχή των χρηστών και όχι σε άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ κύριε Φορσόγκας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας παρουσιάσετε ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο επίσης στον άλλο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας κάνει και αυτό στην ε, παρουσίασή του. Με συγχωρείτε, θα ακολουθήσει ο κύριος Ρομπέρα από τον Όσα. So, um, as of introduction, um, Θα ξεκινήσουμε μία εισαγωγή. Θα σας παρουσιάσω λίγο τα όσα έχουμε κάνει στα πλαίσια του πλαισίου για τα BEPS στον ΩΣΑ, δηλαδή για τις προκλήσεις που δημιουργεί τη φορολόγηση ή η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός κόσμος. Ξεκινήσαμε με το πρώτο ε, BEPS, γνωρίζοντας πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχαμε μια σειρά από φορολογικά σκάνδαλα που μας οδήγησαν στην προσπάθεια δημιουργίας φορολογικού ε, πλαισίου για τις πολύ ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις. Το 2014 λοιπόν η πρώτη προσπάθεια με πρώτη έκθεση που υποβλήθηκε το 2015 και η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε πως δεν έχει κλείσει, πως χρειάζεται να δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φοροαποφυγή και έχουμε ε, μία νέα ομάδα οργασίας η οποία ονομάζεται Task Force για την ψηφιακή οικονομία με νέα εντολή το 2016 και 2017 στα πλαίσια του ε, πλαισίου για τα BEPS ε που είναι το νέο βήμα στο οποίο παρακολουθούμε και εποπτεύουμε το πώς ε, τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται. Και πρέπει να σας πω πως εδώ έχουμε πια σήμερα πάνω από 117 μέλη τα οποία εργάζονται σε ισότιμη βάση. Στα πλαίσια αυτής της νέας εντολής, η Task Force συνέχισε τις προσπάθειές της με μία προθεσμία η οποία αρχικά είχε μπει για το 2020, μετακινήθηκε και είπαμε ότι θα βρούμε κάποιες λύσεις για τα δυσεπίλητα πρόβλημα, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε σε μία ενδιάμεση έκθεση τον Μάρτιο του 2018. Και θα σας παρουσιάσω εντάχει κάποια από τα συμπεράσματα. Πριν όμως μπούμε σε αυτά, θα ήταν χρήσιμο να μπούμε στην πρώτη έκθεση του 2015 για τα BEPS, στα συμπεράσματα εκεί και στα ευρήματα τα οποία δημιούργησαν το έδαφος στο οποίο τώρα εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο. Το πρώτο εύρημα είναι πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κλάδος οικονομίας που να είναι η ψηφιακή οικονομία. Είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης ολόκληρης της οικονομίας, οπότε δεν μπορούμε να περιχαρακώσουμε ε, κάποιες επιχειρήσεις και κλάδους λέγοντας πως φορολογικά αυτά θεωρούνται ψηφιακή οικονομία. Δεύτερον, όταν εξετάζουμε τα διάφορα πλαίσια που δημιούργησαν όλες οι υψηλά ψηφιοποιημένες εταιρείε, διαπιστώσαμε πως οι τεχνικές που χρησιμοποιούν λογιστικά κτλ. είναι αρκετά διαφορετικές ε, από αυτές που έχουν οι άλλες μία ψηφιοποιημένη εταιρείε. Παρ' όλα αυτά έχουν και πάρα πολλά κοινά στοιχεία και αυτό αποτελεί την κοινή βάση κρίσης για τα BEPS και είπαμε ότι στην πρώτη ε, έκθεση για την ε, ψηφιακή οικονομία με το πρόγραμμα πλαίσιο όπου μιλάμε για την ψηφιακή μεταμόρφωση και την ψηφιοποίηση, τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Δηλαδή, τότε καταλήξαμε στην παραδοχή πως η ψηφιοποίηση και τα σχετικά ε, χαρακτηριστικά τα οποία παρουσίασε προηγούμενος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η μεγάλη ε, ε, εξάρτηση από τα άϊλα, η χρήση και η εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όλα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ δεν δημιουργούν θέματα BEPS, ουσιαστικά οξύνουν κάποια από τα προβλήματα αυτών, ε, ε, κυρίως ε, λόγω φορολογικών τακτικών που ακολουθούνται έτσι ώστε να αποφεύγουν τη φορολόγηση. Είπαμε λοιπόν πως υπάρχουν κάποια, κάποιες προκλήσεις φορολογικές που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής και των μέτρων, αλλά θέματα που εμπίπτουν στην ίδια τη φύση αυτών των επιχειρηματικών μοντέλων, δεν είναι τόσο ηθικά ζητήματα, αλλά κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία αναρωτιόμαστε αν το τρέχον φορολογικό πλαίσιο για άμεση και ήμιση φορολογία θεωρείται ακόμα ικανό. Και είπαμε πως αυτές οι βασικές προκλήσεις θα πρέπει να απαριθμηθούν, να περιγραφούν ε, και για την άμεση αλλά και για την έμεση φορολόγηση. Για την έμεση όπως ξέρετε και εσείς έχουν ήδη προκριθεί κάποιες λύσεις και είχαν σχεδιαστεί από τότε και σήμερα έχουμε πια για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, κάποιες παγκόσμιες λύσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές από πολλά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, λόγω των σχετικών με τον ΦΠΑ ε, οδηγής... αλλά και άλλες 60 χώρες που σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζουν τις παγκόσμιες αυτές ε, λύσεις για το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ξέρω πως τα γνωρίζετε. Εδώ το πρόβλημα είναι η αποτελεσματική συλλογή στη χώρα κατανάλωσης όταν ο πάροχος υπηρεσίας ή ψηφιακού προϊόντος δεν βρίσκεται, ε, δεν έχει φυσική παρουσία στη χώρα κατανάλωσης. Για την άμεση φορολόγηση και το κομμάτι εκεί, αντιμετωπίσαμε το εξή πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί. Και νομίζω ότι αυτά εξήγησε και προηγουμένως η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για κατανομή κερδών, για τον έξους, για τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε σχήματα τα οποία εντάσσονται στο τρέχον φορολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, ποιος έχει το δικαίωμα φορολόγησης και ποιος με τα δικαιώματα αυτά. Αυτό δεν ήταν έντολη της ε, Task Force, αλλά ε, θέλαμε να δούμε το θέμα αυτό τη κατανομής δικαιωμάτων φορολόγησης και συμφωνήσαμε πως χρειάζεται παραπάνω δουλειά στους κλάδους αυτούς, έτσι ώστε ε, αργότερα να δοθεί και εκεί μια λύση. Εδώ δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, αλλά η συμφωνία ήταν να συνεχιστούν οι προσπάθειες. has been adopted since uh, BEPS package was Έχουμε και μία νέα εντολή για το πακέτο. Και εδώ τα κομβικά σημεία σχετίζονται με τις ευρύτερες ε, προκλήσεις στην άμεση φορολόγηση που επαναλαμβάνω κατά τη διάρκεια του Project PEPS δεν βρήκαν μια λύση. Και για να έχουμε μια συνενετική προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Το πιο σημαντικό ήταν καταρχήν να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για το τι συμβαίνει και μετά να παρακολουθήσουμε όποιες σχετικές εξελίσει έχουμε και που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, όπως επίσης και με τον τρόπο από τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών που φέραμε σε πέρας και που βρίσκονται στην ενδιάμεση έκθεση, δηλαδή εδώ γίνεται μια ανάλυση των επιχειρηματικών μοντέλων γιατί είναι μοντέλα τα οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ψηφιοποιημένα και επίσης παρακολουθήσαμε την εφαρμογή των BEPS και τις επιπτώσεις που έχει σε ε, εισρωές, εκροές, στα επιχειρηματικά μοντέλα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα ε, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το κομμάτι της φόρου αποφυγής και βέβαια να παρακολουθήσουμε τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη με την ψηφιοποίηση, με τις προκλήσεις σε φορολογικό επίπεδο, ξέρετε πως αρκετά κράτη έχουν υποβάλει προτάσεις σαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό το, η πρόκληση της ψηφιοποίησης. Και αρκετά κράτη, όπως η Ινδία για παράδειγμα, έχει την, ε, ε, την εξισωτική εισφορά ε, που ισχύει. Και ο στόχος είναι να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση εμείς για το ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα κάποιου πρόοδου έτσι ώστε να επιτευχθεί συνένεση για μια μακροπρόθεσμη λύση. Ε, σημαντικό σημείο σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση από φέτος το Μάρτιο ήταν η δημόσια διαβούλευση που οργανώθηκε στην Καλιφόρνια με μεγάλη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους από πολύ διαφορετικές ε, προελεύσεις. Και βέβαια, όλη η διαδικασία αυτή και η νέα εντολή και τα παλαιότερα BEPS έχουν ε, ε, γίνει υπό την αιγίδα του ε, πλαισίου SDG20 που εγκρίνει τις διάφορες φάσεις των ευρημάτων και ανανεώνει τις εντολές της Task για την ψηφιακή οικονομία. Η πιο πρόσφατη έγκριση είναι αυτή της ενδιάμεσης έκθεσης του Μαρτίου του 2018 η, η Προεδρία Αργεντινής. Περνάμε τώρα στην ενδιάμεση έκθεση. Εδώ έχουμε οκτώ κεφάλαια που καλύπτουν πάρα πολλά διαφορετικά θέματα και πιστεύω πως ίσως εδώ το πιο σημαντικό είναι να τονίσουμε το τι έχουμε κάνει ήδη για τις ευρύτερες φορολογικές προκλήσεις. Και βλέπετε εδώ τα διάφορα θέματα που έχουμε εντάξει στην ενδιάμεση έκθεση και αν κοιτάξετε δεξιά, που είναι θέματα φορολογικής πολιτικής, θα διαπιστώσετε πως καταρχήν σημειώθηκε πρόοδος στη διερεύνηση των προκλήσεων αυτών και των συνεπειών των βασικών χαρακτηριστικών της α, ψηφιοποίησης για το φόρο εισοδήματος. Έχουμε την εξάρτηση από τα ΆΙΛΑ, την συμμετοχή χρηστών, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προεκτάσεις που επηρεάζουν τα φορολογικά και τα κράτη έχουν δει το θέμα αναγνωρίζοντας πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι διαφορετικές οι απόψεις για το τι θα πρέπει να γίνει με την ψηφιοποίηση και με τα διάφορα στοιχεία πληροφορικής που χρειάζεται κάθε διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο για να, για να λειτουργήσει. Οι θέσει των κρατών, όπως βλέπετε εδώ, για τις ψηφιακές επιπτώσεις για τη φορολογία εισοδήματος, είναι αυτές που εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες και έχουμε τρεις κατηγορίες κρατών που εμείς εντοπίσαμε. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτές οι χώρες που θεωρούν πως το πρόβλημα σχετίζεται με ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης που είναι η χρήση, η συμμετοχή των χρηστών. Και εδώ χρειάζεται στοχευμένες αλλαγές ε, στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο, αλλά το αφήνουν εκεί μια δεύτερη ομάδα κρατών που θεωρεί πως η ψηφιοποίηση είναι ένα σύμπτωμα απλώς ενός μεγαλύτερου προβλήματος που το προκαλεί η παγκοσμιοποίηση και κάποιες από τις βασικές αρχές της τρέχουσας φορολογικής πολιτικής δεν είναι ε, αρκετά εξελιγμένη για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις δεν περιορίζονται στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να δοθούν αποκρίσεις σε ευρύτερα προβλήματα, οπότε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί γενικότερα σε όλη την οικονομία. Και τρίτη κατηγορία κρατών που θεωρεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που να σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και όταν εφαρμοστούν τα BEPS θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Εδώ είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση από όλα τα κράτη στο πλαίσιο ανεξάρτητα με το σε ποια ομάδα κρατών που περιέγραψαν ανήκουν και έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να βρουν μια μακρόπρόθεσμη λύση που θα ε, αλλάξει και τους κανόνες κατανομής ε, κερδών αλλά και τα όσα σχετίζονται με τον έξους. Και θα κλείσω λέγοντας πως νομίζω πως μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το κατά πόσο είναι βιώσιμη η πρόοδος στο κλάδο αυτό γιατί θεωρούμε πως έχουμε την τελική προθεσμία του 2020 και μία από τις βασικές χώρες που, θα είμαι ειλικρινής, ε, προσπαθούσε να μπλοκάρει ε, την πρόοδο στις συζητήσεις αυτές, γιατί ε, διαφωνεί με την διάγνωση ήδη που κάνουμε και για τον τρόπο που βλέπουμε την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση, ή είπα, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει στο να συζητηθούν τα θέματα αυτά και έχει δεσμευθεί μαζί με τις υπόλοιπε χώρες, ζητώντας να γίνει μια τροποποίηση στη, στους τρέχοντες κατε, κανόνες κατανομής κερδών και ενέξους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Και εδώ, στην τελευταία διαφάνεια, εντοπίζουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα σε επίπεδο task force. Και ποιο είναι το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα εργασίας για να πετύχουμε συνένεση για μακροπρόθεσμη λύση, Κάποιες τεχνικές λοιπόν εργασίες για το τι, θα πρέπει, τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η μακροπρόθεσμη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. for questions. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρομπέρ για την παρουσίαση της θέσης του ΩΣΑ. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα γίνουν τώρα οι ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν διάρκεια πέραν του ενός λεπτού. Και θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την παρουσίαση αυτή. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την ακρόαση που είχαμε στην ΕΚΟΝ Πιστεύω ότι εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μία πιο δίκαιη κατανομή της φορολόγησης. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να δημιουργηθεί διπλή φορολόγηση. Είτε αν θέλετε την φορολόγηση ενός υπάρχοντος ε, κέρδος το οποίο έχει ήδη φορολογηθεί, υπάρχει αυτή η, αυτός ο κίνδυνος και βάσει ποιων στοιχείων θα γίνεται η εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ψηφιακή οικονομία, αλλά και παραδείγματος χάρη ε, τις πωλήσει ε, εξ και άλλου είδους εμπορικές συναλλαγές και όχι μόνο την ψηφιακή οικονομία. Συμφωνείτε? Και όσον αφορά την κατανομή του κέρδους είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σωστή κατανομή του κόστους. Είναι ίσως λίγο πιο γενική η ερώτησή μου. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε το κόστος και τη βάση κόστους για αυτήν την ε, νέα ε, ίδρυση, αν θέλετε, φορολογικής βάσης. Ευχαριστώ. Κύριε Ρομπέρ, θέλετε να απαντήσετε. Μπορώ να σχολιάσω το δεύτερο σημείο της παρέμβασής σας. Νομίζω ότι όσον αφορά τη διάβρωση της ε, φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και που θεωρούν ότι ουσιαστικά η ψηφιακή οικονομία αυτό που κάνει είναι ότι υπερβάλλει και μεγιστοποιεί υπάρχοντα προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό, μια σημαντική ομάδα ε, χωρών που κάνει αυτή τη διαπίστωση. Αν συμφωνείτε, αν και εσείς κάνετε αυτή τη διάγνωση, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν λύσεις βραχυπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες. Καταρχήν, εντοπισμός των συγκεκριμένων ε, χαρακτηριστικών μιας αγοράς, χαρακτηριστικά που αφορούν μια χώρα ή μια αγορά, συγκεκριμένοι τρόποι για να υπάρξει τροποποίηση του υπάρχοντος πλαισίου και μέτρα για να φτάσουμε σε μια πιο δική κατανομή ε, της ε, φορολογίας και τέλος να εντοπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος, του σημερινού συστήματος, έτσι ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη φορολόγηση στο μέλλον και να πάψουν να υπάρχουν τα κενά και οι αδυναμίες που σήμερα επιτρέπουν αυτές ε, τις ε, στρεβλώσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε πρόσβαση σε μια αγορά, να μπούμε σε μια αγορά και ενδεχομένως να συζητήσουμε τις διάφορες ε, εναλλακτικές λύσεις και λύσεις βραχυπρόθεσμες ή πιο μακροπρόθεσμες. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα που κάνατε. Εγώ συμφωνώ. Δεν θέλουμε να φορολογήσουμε περισσότερο, αλλά διαφορετικά και αυτό ουσιαστικά με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο, δηλαδή να αλλάξουμε τους υπάρχοντες κανόνες έτσι ώστε να ενσωματωθεί η νέα ψηφιακή οικονομία και τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και με τα μεσοπρόθεσμα, τα προσωρινά αυτά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί. Θέλουμε να κανονίσουμε με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο καταρχήν το γενικότερο πλαίσιο, τις αγορές που ε, σήμερα λειτουργούν, τις εταιρείες που έχουν φυσική παρουσία, δεν έχουν φυσική παρουσία, δημιουργούν κέρδος και να βασίσουμε την φορολογία και στη φυσική παρουσία αλλά και στην ε, φορολόγηση των κερδών. Ε, και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι γιατί θα πρέπει εδώ να ισχύουν οι κανόνες αυτοί και στις ε, εσωτερικές αγορές, στις εθνικές αγορές. Όπως ξέρετε, η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτό, de facto, οδηγεί όμως σε διακρίσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει εδώ να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, εθνικές αγορές, τις εσωτερικές αγορές, έτσι ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις, να επιτρέψουμε δηλαδή στις ε, ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις αλλά και σε παγκόσμιους ομίλους να συνυπολογίσουν όλες τις δραστηριότητες τους εντός και εκτός των συγκεκριμένων αγορών που φορολογούνται. Το θέμα τώρα της ύπαρξης των αξιόπιστων στοιχείων, βεβαίως εδώ όλες οι χώρες δεν επιτρέπουν την επιβολή αυτών των κανόνων και το θέμα της επιβολής ενός ευρωπαϊκού φόρου, μιας ευρωπαϊκής φορολογίας σε μια μη ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Μια αμερικανική εταιρεία, ινδική, κινέζικη εταιρεία. Θα πρέπει ουσιαστικά να είναι κατανοητό στον Ευρωπαίο καταναλωτή ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλουν των ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία τύπου one-stop shop, μια διαδικασία διαφανής και απλή, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να μην δυσκολεύουν την ε, εισπράξη του φόρου την κατανόηση των κανόνων και σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά τα οποία διαφεύγουν πάνω από 750 εκατομμύρια συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θέστε κάποιες ερωτήσεις. Συνεισηγητής για το S&D. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Από το τελευταίο ερώτημα, για να είμαι ακριβής, Πολύ συχνά ακούγεται το εξή επιχείρημα. Έχουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ότι υπάρχει παράκαμψη της φορολογήσεως από τι ψηφιακέ εταιρείε που είναι εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσης, εδρεύουν εκτό, αλλά δραστηριοποιούνται στην ενία αγορά. Μπορείτε να μα πείτε ποια είναι η κατάσταση με το Facebook να συνεχίσει να, πουλεί, να πουλά τι υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την θέσπιση αυτών των διατάξεων χωρίς να υπόκειται στην ψηφιακή φορολόγηση. Νομίζω το απαντήσατε, αλλά είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά. Άλλο ένα επιχείρημα που συχνά ακούγεται κατά της ψηφιακής φορολογήσεως. Τι γίνεται με τις μη ψηφιακές εταιρείες. Δηλαδή η αρχή της φορολόγησης στον χώρο που παρέχεται υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχει μία ψηφιακή παρουσία. Μπορείτε να μας πείτε αν η προτασή της φορολόγησης ψηφιακής υπηρεσίας θα ισχύει και για παραδοσιακές εταιρείες μη ψηφιακές, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες ή αυτές που παράγουν άλλα φυσικά προϊόντα, παιχνίδια, φερρυπίν ή ενδύματα. Και τέλος προς τον ΩΣΑ, τον κύριο Γομπέα. Ήσασταν πολύ αισιόδοξο όσον αφορά την κοινή δράση και τη συμφωνία και συνένεση μεταξύ χωρών του ΟΣΑ μέχρι το 2020. Πού βασίζεται η αισιοδοξία σας. Ε, ελπίζω να έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προστατεύσει την κυριότητα τη ενίας αγοράς, να εξασφαλίζει θεμητού όρου, ισότιμού όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφευθεί η διάβρωση της φορολογητέας βάσεως μέσω των προτάσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως το συζητάτε αυτό και στα πλαίσια του, των συζητήσεων του ΟΣΑ, της προσωρινής διατάξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω την τελευταία ερώτηση. Πού θα εφαρμοστεί αυτή η φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών. Θεμελιώδες θέμα δεν είναι φόρος επί εταιριών συγκεκριμένων ή επί ομίλου εταιριών, δεν είναι φόρος που αφορά συγκεκριμένο τομέα, ούτε φόρος επί ψηφιακών εταιριών. Όπως είπατε σωστά, μπορεί να έχετε και παραδοσιακή εταιρεία που παρέχει κάποιες υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο του DST. Είναι ένας φόρος ο DST που πρέπει να καταβάλλεται από φορολογούμενα πρόσωπα βάση κριτηρίων και που παρέχουν κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες καθορίζονται καλά στην οδηγία. Διαφημιστικές υπηρεσίες, μια μετάφραση πώληση στοιχείων. Αν πάρουμε μια φαρμακευτική εταιρεία, Φερρυπίν, παραδοσιακή εταιρεία, που πολλή στοιχεία, όχι οποιαδήποτε στοιχεία, στοιχεία που καθορίζονται σαφώς από την ομοθεσία που παράγονται από τους χρήστες μέσω ψηφιακών πλατφορμών κλπ. Αυτή η εταιρεία εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογή του DST. Για την πρώτη ερώτηση, δεν την έπιασα καλά. Δεν κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ της δικής σας ερωτήσεως και του προηγούμενου Ευρωβουλευτού. Πώς θα παρακάμπτουν οι εταιρείε ενδεχομένως τη φορολόγηση. Ο κίνδυνος είναι ελάχιστος και δεν είναι χειρότερος από τη δυνατότητα που η ίδια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρακάψει τον φόρο που ήδη έχει καθοριστεί τώρα, που ισχύει τώρα. Οι φορολογικές δικαιοδοσίες πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό για να καλύπτουν αυτούς τους κινδύνους και να ελαχιστοποιούν τους εν λόγω κινδύνους και αυτό το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ, Όσα. a few words on the um, Θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα του κατά πόσο είμαστε αισιόδοξοι για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στα πλαίσια του All-Inclusive Framework και κυρίως στο ότι διαπιστώνουμε να υπάρχει ε, μία νέα δυναμική. Έχω ξεκινήσει με το project αυτό το 2013 και το παρακολουθώ έκτοτε, δηλαδή έχουν πέρασει πάνω από πέντε χρόνια και πρέπει να σου πω ότι η δυναμική άλλαξε στην Task Force. Οι ισορροπίες άλλαξαν και δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, δεδομένης της νέα ε, θέση που έχουν λάβει κάποια κράτη. Για τις ε, μονομερείς δράσεις και κυρίως για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό φόρο υπηρεσίας, αν δείτε τα δικά μας μέλη δεν υπάρχει συνένεση για το κατά πόσο χρειάζεται μια άμεση και μονομερής δράση στο σημείο αυτά. Και δεν μοιάζει να είναι πιεστική αυτή η ανάγκη. Και τώρα, εκ μέρους του ΩΣΑ, να σας πω πως θεωρούμε πως το δικό μας DNA βρίσκεται το να πετυχαίνουμε πολυμερείς συνενετικές λύσεις. Οπότε έχουμε μία φυσική αποστροφή προς τις μονομερείς και μη συντονισμένες μεταξύ τους δράσης. Πολλές από τις χώρες που ανήκουν στη Task Force, εκτός από αυτές που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν με συμπάθεια και κατανόηση τις πιέσεις τις οποίες ε, αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και άλλα κράτη στον κόσμο που ε, αισθάνονται την ανάγκη και πιέζονται να αναλάβουν άμεση δράση και στην διάμεση, διάμεση έκθεση αυτό αναγράφεται. Βεβαίως ε, τα κράτη επιτρέπονται, επιτρέπεται στα πλαίσια του εσωτερικού δικαίου να ε, νομοθετούν όπως το επιθυμούν, αρκεί να είναι εντάξει με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Η μόνη βασική γραμμή στον ΩΣΑ είναι πως οποιαδήποτε μονομερής δράση αναλαμβάνει μια χώρα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο που δεν θα υποσκάφτει την πρόοδο την οποία εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε τη στιγμή που σχεδιάζουμε μια μακροπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν έχουμε τις, ε, ε, την ευκαιρία να μιλήσουν και οι συνεισηγητές από την ΕΚΟΝ, Νταρίους. Ναι. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχήν. Τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργήσει η διάκριση μεταξύ ψηφιακών υπηρεσιών που θα φορολογούνται και άλλων ψηφιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν κάποια κράτη. Είναι εύκολο να γίνει αυτό σε κάθε περίπτωση και με σαφήνεια να ε, οριοθετηθεί δηλαδή έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαιές ζώνες όπου κανείς δεν θα γνωρίζει ποια είναι η φορολογητέα η υπηρεσία και ποια όχι. Για μένα δεν είναι τόσο σαφές γιατί οι ορισμοί ακόμα είναι γενικόλογοι. Και σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως οι εθνικές φορολογικές αρχές είναι έτοιμες να κάνουν αυτή τη διάκριση και να μετρήσουν αυτές τις φορολογητές ψηφιακές υπηρεσίες. Είστε πεπισμένους πως έχουν τη δυνατότητα να το αξιολογήσουν αυτό και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις προτάσεις. Επίσης έχω μία ερώτηση και στρέφομαι προς τον ΩΣΑ είναι λίγο συνέχεια τη προηγούμενη ε, ερώτηση. Κάποια κράτη στον ΩΣΑ είναι κατά αυτής της φορολογίας, ε, τουλάχιστον είναι κατά τη γενικότερη ε, έννοια του ψηφιακού φόρου. Γιατί λοιπόν είναι εναντίον, ποια είναι τα επιχειρηματά τους και εσεί είστε ακόμα πεπισμένους πω θα βρείτε μια λύση συμβιβαστική μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια για να έχουμε μια μαγκόσμια λύση. Εάν ναι, τι είδους επιχειρήματα η τακτική προτείνετε για να πείσετε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να σας ακούσουν και δεν θέλουν καθόλου να σκεφτούν αυτή τη ε, δυνατότητα. Επίσης, σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η μονομερής δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εγώ στηρίζω, βοηθά προς την εξέβρεση μιας παγκόσμιας λύσης γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αυτή τη δράση με τούτο το εργαλείο μόνη της. Πιστεύετε πως αυτό παρακινεί τα άλλα κράτη προς μια κοινή λύση. Ή τα προκαλεί να αντισταθούν. Τι πιστεύετε. Είστε υπέρ των όσων κάνουμε εδώ. Αυτό τον οποίο ξεκινήσαμε μέσω της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω των δικών μας εκθέσεων. Ευχαριστώ πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yeah, thank you for your question. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Η διάκριση μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, όπως τις περιγράφουμε και στην οδηγία, καταρχήν πιστεύω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ στοχευμένη οδηγία που καλύπτει μόνο τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες και ουσιαστικά στην πράξη δεν έχει επιπτώσεις αυτό όσον αφορά την εφαρμογή του νομοθετικού αυτού κειμένου. Και βεβαίως ε, όσο λιγότερες ε, υπηρεσίες συμπεριλαμβάνει ένα κείμενο, τόσο πιο εύκολη είναι η εφαρμογή του. Και όσο περισσότερες, τόσο πιο πολλά προβλήματα προκύπτουν ως προς την εφαρμογή. Βεβαίως καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, όχι μόνο από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και από μέρους μεμονωμένων κρατών. Μπορούμε να διευκρινίσουμε και οι ερωτήσεις σας μας βοηθούν ποιες φορολογικές υπηρεσίες ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Είμαστε ανοιχτοί και δεχόμαστε σχόλια από μέρους σας εάν αυτά οδηγούν σε περισσότερη αποσαφήνιση και διευκρίνηση του κειμένου. Όσον αφορά τους ορισμούς, όπως σε κάθε νομικό κείμενο, ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολύ συγκεκριμένες έννοιες όπως οι εξαιρέσεις, τι παραδείγματο χάρη εξαιρείται, σε ποιες υπηρεσίες επιβάλλεται ΦΠΑ ή άλλη φορολόγηση για να μην γίνονται ε, λάθη και διακρίσεις. Και βεβαίως ε, έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος, ε, η εκτίμηση και να συμμορφωθούν με τα κείμενα όταν θα ψηφιστούν. Όσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το πρώτο σημείο που αφορά το DST, γιατί κάποιες χώρες, παραδείγματο χάρη, συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες όσον αφορά την υιοθέτηση ένας από τους λόγους θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχουν ε, οικονομικές τρευλώσεις που ουσιαστικά απορρέουν από τέτοια μέτρα. Η κάθε μονομερής ε, δράση, η κάθε εθνική δραστηριότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται, να συνάδει με τις διεθνείς ε, αρχές που φυσικά συμπεριλαμβάνουν την αρχή της μη διάκρισης και φυσικά και όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι αν θέλετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει περιθώριο ελιγμού. Η κάθε χώρα μπορεί να σχεδιάσει τα δικά της μέτρα, τα οποία να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στη δικέ στις δικές της ε, ιδιαιτερότητες, ε, στα χαρακτηριστικά της δικής της οικονομία. Κάτι άλλο που ακούσαμε από άλλες χώρες είναι ότι οι μακροπρόθεσμες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν με προθεσμία το 2020 και το ερώτημα αν ε, αξίζει να υιοθετηθούν σήμερα προσωρινά μέτρα, γιατί το 2020 είναι πραγματικά και βάση των ε, διαδικασιών του ΟΣΑ, αλλά και οι νομοθετικές διαδικασίες των κρατών μελών είναι τόσο χρονοβόρες που το 2020 είναι αύριο το πρωί. Είναι πάρα πολύ μικρή ε, στενή προθεσμία. Υπάρχει λοιπόν λόγος προσωρινών μέτρων, αλλά όσον αφορά μονομερή άμεση δράση, τύπου DST ή άλλα μέτρα σε αντιπαράθεση με μακροπρόθεσμες λύσεις και μέτρα, Σίγουρα κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των μακροπρόθεσμων μέτρων τα έχουμε ήδη συζητήσει, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει μια ρήτρα προθεσμίας ε, ή ημερομηνία λήξης, όσον αφορά δηλαδή την λήξη αυτών των μέτρων, σε περίπτωση που τελικά υιοθετηθούν, συμφωνηθούν ε, μακροπρόθεσμες λύσεις σε διεθνές επίπεδο. Κάποιες χώρες μπορεί να θεωρήσουν ότι η πρόταση για υιοθέτηση μονομερών μέτρων μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο, έτσι ώστε να πιεστούν άλλες χώρες για να υπάρξει συμβιβασμός και για να υπάρξει σύγκληση, μέτρα σύγκλησης και βήματα προς την κοινή κατεύθυνση. Αυτό για μένα είναι κάτι το πολιτικό, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ευχαριστώ. Έχουμε οκτώ ομιλητέ που αντιπροσωπεύουν πολιτικές ομάδες. Πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των ερωτήσεων και να βραχύνουμε στο τετράλεπτο το χρόνο παρέμβασης εκτός μικροφώνου συζήτησης. some... Και για κάποιους άλλους υπήρχε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που διατέθη, αλλά ήταν συνεισηγητές. Ήταν κάτι διαφορετικό. Τέλο πάντων. Ότμαρ Κάρας για το ΕΛΚ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Δεν μιλάμε μόνο για θέματα που αφορούν, ε, αν θέλετε, επιχειρήσεις ε, με ύποπτες πρακτικές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο σημαίνει και εντός. Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ξέρετε πολύ καλά ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο ΕΚΟΦΗΝ συζητήθηκαν τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σίγουρα θα πρέπει να ξαναδεί τον κανόνα της ομοφωνίας για τέτοιου είδους θέματα, κάτι που πραγματικά εμποδίζει αποτελεσματικές αποφάσεις. Επίσης το θέμα της α, κακής θα έλεγα οριοθέτησης του ψηφιακού και μη ψηφιακού κόσμου στην οικονομία. Θα πρέπει να δούμε λίγο και τα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Για μένα το ιδανικό θα ήταν αυτά να σε ένα μείγμα, γιατί εδώ μιλάμε για το 3%, μιλάμε για δισεκατομμύρια, για το 3% της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έσοδα, οι ίδιοι πόροι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας. Κάναμε μια πρόταση. Αναφέρεστε στον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών και τα προσωρινά μέτρα. Κάναμε πρόταση βάσει του άρθρο 113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί ομοφωνία. Αυτό είναι το ενδεχόμενο που επεξεργαζόμαστε. Για τη δεύτερη ερώτηση. Ψηφιακές υπηρεσίες, μη ψηφιακές, διάκριση. Τίθεται στο θέμα της συζητήσεως. Τι αποτελεί ψηφιακή υπηρεσία, τι όχι. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να μείνουμε εκτός αυτής της συζητήσεως. Πώς? Καθορίζοντας κάποιες υπηρεσίες συγκεκριμένες και τα χαρακτηριστικά αυτών. αυξήσαμε την ασφάλεια δικαίου ότι ο τρόπος για τις εφοριακές αρχές και τι επιχειρήσει όσον αφορά την ταξινόμηση δραστηριοτήτων στον πραγματικό κόσμο. και ποιε δραστηριότητε είναι αυτέ που πρέπει να φορολογηθούν από τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Ζητώ συγγνώμη αν δεν απαντώ έτσι στην ερώτησή σα, πείτε το μου. Μετά, η δυνατότητα που υπάρχει να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από ψηφιακό, το, φόρο ψηφιακών υπηρεσιών για τους ιδίους πόρους. Στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει το ψηφιακό φόρο και το σχετικό πακέτο γινόταν μενία αυτής της δυνατότητας. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί εκτενώς το συγκεκριμένο θέμα που θέσατε. Mrs. Κυρία Σλάιν, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάλεξε το 3% για αυτό το προσωρινό ψηφιακό φόρο. Μετά από σεχτική ανάλυση διαφόρων παραγόντων, λέει, και αντιχτύπου βάρους φορολόγησης των επιχειρήσεων με διαφορετικά περιθώρια κέρδους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε περισσότερο αυτό που προανέφερα, που είπατε. Άλλη ερώτηση. Πόσες εταιρείε όλο τον κόσμο είδα τα στοιχεία που αναφέρετε στην παρουσίασή σας. Έχετε κάποια ιδέα πόσες εταιρείε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φορολογήσιμα πρόσωπα σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 4. Τελευταία ερώτηση. Αυτό πώς ταιριάζει με την απαιτούμενη διαθροτική απάντηση στην οδηγία CCTB. Μήπως έτσι καθυστερεί η, έγκριση του CCTB. Και από αυτού το Κοινοβούλιο επανειλημμένα μεγάλη πλειοψηφία θεώρησε και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη Καταρχάς, διότι η ομάδα που εξεργάστηκε το θέμα είναι αρκετά πολυμελής. Δεν μείνατε δυστυχώς με τους οικονομολόγους της ομάδας και συγχωρήστε μας για τις βασικές εξηγήσεις που θα σας δώσουμε. Με τα χαράς να διαβιβάσουμε ε, τυχόν γραπτές ερωτήσεις αργότερα και στο βαθμό του δυνατού να διευκρινίσουμε τις απορίες. Το 3% αυτό αποφασίστηκε ούτως ώστε να εξισορροπηθεί η ανάγκη συλλογής εισοδημάτων για να αντισταθμιστούν οι δαπάνες στην εφαρμογή του μέτρου και απ' την άλλη παραδεχόμενοι το ότι αυτός ο συμπληρωματικός φόρος πιθανότατα θα δημιουργούσε στρεβλώσεις στην περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείε που πληρώνουν τον ψηφιακό φόρο ε, ταυτόχρονα υπόκεινται και σε φόρο ε, εταιρικό σε ένα Διάφορα περιθώρια λήφθησαν υπόψη και οι, οι, εταιρείε που θα υποστούν τη διπλή φορολόγηση αυτή είναι κάτι που έχει υπολογιστεί. Ποσοστό πάνω από 3% οδηγούσε σε επίπεδα φορολόγησης που θεωρήθηκαν ότι παρεμποδίζουν και παρενοχλούν σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα των εταιριών αυτών. Ενώ χαμηλότερος φόρος, χαμηλότερο ποσοστό φορολόγησης δεν εξασφάλιζε την οικονομική βιωσιμότητα του φόρου αυτού καθεαυτού. Γι' αυτό 3% κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο προαναφερθησών πτυχών που χρειαζόταν εξισορρόπηση. Για δεύτερη ερώτηση, εκτιμούμε ότι περίπου 180 με 200 εταιρείε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να υποστούν αυτό το φόρο του ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι εταιρείε που ξεπερνούν τα δύο όρια και που παρέχουν φορολογητέ υπηρεσίε. Και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο όσον αφορά το CCTB. Βάσει τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το CCTB δεν εφαρμόζεται στι εταιρείε διότι υπάρχει πρέπει να έχουν τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα για να, μπουν σε αυτό το πλαίσιο εταιρείε. Αν εγκριθεί το CCCTB και πάλι χαζόμαστε κανόνες για άλλες εταιρείε που δεν υπόκειται στους κανόνες του CCCTB. Τούτου λεκθέντος αναγνωρίζουμε πράγματι ότι οι προτάσεις για την κοινή βάση και το CCCTB θα πρέπει να προσαρμοστούν εν ευθέτω χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τις στοιχές της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την ψηφιακή παρουσία και θα πρέπει να προσαρμόσουμε δεόντως τους τύπους περί Και το Ευρωκοινοβούλιο έκανε ενδιαφέρουσε ε, προτάσεις σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σλάιν γιατί κάνατε πολύ καλή ερώτηση σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ε, από τους φιλελεύθερου ο συνάδελφο, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη τύχη και δεν καταφέραμε εύκολα να βρούμε βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ε, σε θέματα φορολογικά. Γιατί λοιπόν πιστεύετε πως ε, αυτή τη στιγμή ο φόρος της υπηρεσίας, ψηφιακής υπηρεσίας θα έχει καλύτερη τύχη. Τι θα γίνει, θα έχουμε την ίδια τύχη με τον φορό για τις ε, συναλλαγές, νομίζω θα χρειαστεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και θα φορολογούμε τα κέρδη ή τον κύκλο εργασιών έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και κάποια κέρδη τα οποία δεν εμφανίζονται. Ε, δεν φοβόσαστε εσείς ε, τι θα γίνει και αν θα πάρουν αντίματρα αυτές οι εταιρείες, οι κολοσσοί, οι αμερικάνικες, οι οποίες είναι οι βασικές που θα φορολογηθούν. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί ο φόρος αυτός της ψηφιακής υπηρεσίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά με πολύ πιεστικές προθεσμίες για να σχεδιάσουμε τρεις προτάσεις και μία πλήρη επιδοσιολογική μελέτη, η οποία να είναι σε τεχνικά ε, στέρεη βάση και αναγνωρίζουμε πως μας έχει ασκηθεί κάποια κριτική, ξέρουμε ποια είναι αυτή, αλλά θέλω να τονίσω πως δεν έχω ακούσει να υπάρχουν σοβαρές εναλλακτικέ λύσεις προτάσεις που εμείς έχουμε καταθέσει. Αυτό πρέπει να το δούμε. Θέλουμε να είναι τεχνικά βάσιμες οι προτάσεις μας, όταν τις καταθέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να λαμβάνουμε υπόψη αφού ακούσουμε οποιασδήποτε λογικές προτάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη ποιότητα σε αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Γιατί δεν κάνουμε φορολόγηση σε κέρδη και σε εισόδημα και κάνουμε ε, προσπάθεια φορολόγηση κύκλου εργασίας ε, δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, αλλά ελήψη μιας ε, παγκόσμιας λύσης, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, θεωρούμε πως μια ευρωπαϊκή αλλαγή των κανόνων ε, για την εταιρική φορολογία, δηλαδή κάτι που συνδυάζει τα έσοδα και το κέρδος και φορολογία αυτά από κοινού, θα είναι η καλύτερη δυνατόν επιλογή. Όμως θα πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικές ουσιαστικές ε, πτυχές του, ε, της φορολογίας επιχειρήσεων. Οπότε, εντωμεταξύ, χρειαζόμαστε κάποια διάμεσα μέτρα ε, τα οποία θα ασκήσουν όσο συζητάμε, θα, θα εφαρμόσουμε όσο συζητάμε τις παγκόσμιες λύσεις. Είπαμε, παγκόσμιος φόρος στις, στον όγκο συναλλαγών και όχι στα κέρδη, γιατί διαφορετικά αν μείνουμε στις φορολόγηση των κερδών θα παραμείνουμε στο ίδιο επιχειρηματικό πλαίσιο φορολογικά επιχειρηματικό πλαίσιο, στο οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε, δίνοντας μια μακροπρόθεσμη λύση. Οπότε, ως ενδιάμεσο μέτρο, προτείνουμε κάτι διαφορετικό και όχι κάτι το οποίο είναι ίδιο και έχει τα ίδια προβλήματα με τους, κανόνε με κανόνες περί φορολογίας επιχειρήσεων που προσπαθούμε να αλλάξουμε σήμερα. Θέλουμε έναν άλλο μηχανισμό, ένα καινούριο μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα πιο πιεστικά κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της δράσης των ψηφιακών επιχειρήσεων που δεν ε, εμπίπτουν στις κατηγορίες της κλασικής φορολογίας ε, επιχειρήσεων. Για την τελευταία ερώτηση για αντίπεινα και αντίμετρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι θα κάνω οι άλλες δικαιοδοσίες. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω πως δεν πρόκειται εδώ για φορολογία ε, πάνω σε επιχειρήσεις, σε ομάδες επιχειρήσεις, σε όμως επιχειρήσεων από συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Είναι φόρος ο οποίος αντιμετωπίζει, όπως είπα, οποιαδήποτε εταιρεία προσφέρει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες από όπου και να προέρχεται και όπου και να είναι εγκατεστημένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευαζολή για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο του ΟΣΑ εάν προσπαθείτε με την έκθεση αυτή να διορθώσετε κάτι το οποίο δεν ε, διορθώνεται. Βλέπουμε από την ε, πρόσφατη παρουσίαση που κάνατε ότι παρόλο τους καινούριους κανόνες BEPS, ε, παρόλη την νέα διακυβέρνηση, παρόλες τους νέους κανόνες για να πλησιώσουν, το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Δαπανίσατε χρήματα, χρόνο, σειρά, προσπάθειες, συναντήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τεράστια κενά στη φορολόγια. Ακόμα και χώρες όπως η Βραζιλία που έχει μονομερείς κανόνες, βλέπουμε και άλλες χώρες δεν υπάρχει σήμερα αποτελεσματικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω τη, και από την Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογία, πέρα από την Γερμανία που αντιτίθεται σε αυτήν την ψηφιακή φορολογία Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα ποιες είναι οι θέσεις των μεν και των δε και ποια είναι η αναμενόμενη εξέλιξη. Ο Μπρινόλομερ πρότεινε αυτήν την ρήτρα λήξης για τα νέα αυτά μέτρα φορολόγησης. Ποια είναι η άποψή σας, ο κύριος Τροπέρε από τον Όσα. Thank you. Um, uh, thank you. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε πρόσφατες ημερομηνίες. Ουσιαστικά αναφερθήκατε και στα τελευταία μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις του ΩΣΑ. Βεβαίως ε, υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αλλά η προσπάθειά μας είναι να υπάρξει σύγκληση τουλάχιστον στους κανόνες για τους εταιρικούς φόρους. Θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Όσον αφορά το σχέδιο BEPS, το G20, μας είχε δώσει μια συγκεκριμένη εντολή BEPS και αποφυγή διπλής φορολόγησης. Και είναι σωστό το πρέπει να το παραδεχτούμε ότι το 2015 όταν υλοποιήθηκαν οι πρώτες αποφάσεις παρατηρήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα και προσπαθήσαμε να αποφύγουμε καταρχήν όπως σας είπα την διπλή φορολόγηση από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξεπεράσαμε και όλα τα θέματα που αφορούν τη φορολογία και τη φορολόγηση εισοδήματος, τα θέματα ανταγωνισμού, τα εργαλεία που σχεδιάσαμε στα πλαίσια του σχεδίου BEPS δεν συμπεριλαμβάνουν καθόλου θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών. Τα θέματα του νέξους της ψηφιακής οικονομίας και τους κανόνες για την κατανομή των κερδών και την φορολόγηση. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες και όσον αφορά τις χώρες προέλευσης, τις χώρες από τις οποίες προέρχεται μία επιχείρηση, εκεί που έχει την έδρα της και εκεί που δραστηριοποιείται και εκεί που δημιουργείται το κέρδος. Το θέμα είναι ότι από τις προσπάθειες και από το σχεδιασμό μας προκύπτουν πολλές διαφορετικές λύσεις. Και οι λύσεις αυτές σαφώς και έχουν σαν σκοπό καταρχήν την μείωση του... Σας έδωσα κάποια παραδείγματα προηγουμένως, αλλά και ένα επιπλέον παράδειγμα. Η αξία που δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη αγορά, το κέρδος που προέρχεται από τη δραστηριότητα αυτή, το φορολογητέο εισόδημα, το κέρδος και αν θέλετε όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού, άιλα, υλικά, Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Σήμερα, επαναλαμβάνω, η εντολή μας δεν είναι να ασχοληθούμε με θέματα φορολογικού ανταγωνισμού, αλλά η οποιαδήποτε λύση υιοθετηθεί θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση και την εξάλληψη τελικά αυτού του φορολογικού ανταγωνισμού. Σας παρακαλώ πολύ, ε, μπορείτε να απαντήσετε για τη θέση της Γερμανίας. Εμείς δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε, δεν είναι θέση μας να εξηγήσουμε τη θέση της Γερμανίας και ποια είναι η λογική που ακολουθείται πίσω από τη θέση αυτή της χώρας. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι ότι τα κράτη-μέλη όλα προσπαθούν ενεργά να συζητήσουν το θέμα για το πώς να λειτουργήσει το σύστημα. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Όσον αφορά τον χρονισμό για την ε, έγκριση αυτού, ε, στο ECOFIN Υπουργοί Οικονομικών έθεσαν σαν όριο το Δεκέμβριο για να επαναξιολογήσουν την κατάσταση και την επιτευχθήσα πρόοδο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα εξακολουθεί η σκληρή προσπάθεια. Θα εξακολουθεί η σκληρή προσπάθεια και θα φτάσουμε, να δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε. Όσον αφορά τη ρήτα σταδιακή ε, παύση, ε, λήξη. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε του νομικού κειμένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπήρχε τέτοια ρήτρα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τη ρήτρα εκπνοή. Αν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα που έχουμε που εμποδίζει το συμβιβασμό, σίγουρα θα βρεθούν λύσει για να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η ρήτρα σταδιακή εκπνοή δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για μια συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η Γκουε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η ψηφιακή φορολόγηση είναι κάτι που παίζει τεράστιο ρόλο στον τύπο, στα μέσα, στη Γερμανία και αυτό δεν αφορά μόνο το ΕΚΟΦΗΝ, αλλά δημοσιεύθηκαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και έγγραφα την προηγούμενη εβδομάδα καθώς και έντυπα από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών με πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις κατά αυτής της ε, ψηφιακής φορολόγησης. Υπάρχει και η θέση των ε, Αυστριακών. Αυτό δεν έχει κάτι να κάνει με την ε, φορολογική δικαιοσύνη και την πιο δίκαιη κατανομή της φορολόγησης των κερδών. Εσείς Πώς βλέπετε, κύριε Ρομπέρ, την ε, δυνατότητα και τις πιθανότητες μια τέτοια πολιτική φορολόγησης να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί. Ξέρω πολύ καλά πως όσα ορίζει την ψηφιακή οικονομία και πώς περιορίζει πολύ συγκεκριμένα τους τρόπους φορολόγησης, φορολόγησης οδήματος, ε, φορολόγηση κερδών, αποφυγή στρέβλωσης ανταγωνισμού και φορολογικού ανταγωνισμού. Εσείς πώς ε, αξιολογείτε την πιθανότητα μιας τέτοιας ε, πολιτικής η οποία μπορεί να υιοθετηθεί από όλους. Ο κ. Ρομπέρ από πλευρά ΣΟΣΑ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικότατος για την ψηφιακή παρουσία. Τι μπορώ να πω ότι η ενδιάμεση έκθεση εντοπίζει αυτή τη διασύνδεση των έξω σαν ένα τμήμα του προβλήματος και γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό για αλλαγές του έξω για να σχετίζεται λιγότερο ή να μην σχετίζεται καθόλου με τις απαιτήσει περί φυσικής παρουσίας. Αυτό που είναι σημαντικό και που μπορεί να διαγνώσει κανείς διαβάζοντας την ενδιάμεση έκθεση είναι ότι υπάρχει αναγνώριση ότι σημαντικό θέμα δεν είναι το, το έξους, η σχέση αυτή, αλλά η κατανομή του κέρδους. Ε, δεν ξέρω πώς θα λάβουμε υπόψη τη παρουσία. Αν δεν υπάρχει κέρδος που μπορεί να καταναμηθεί, να καταλογιστεί σε αυτή την ψηφιακή παρουσία, δεν έχει νόμιμη προσπάθεια. Γι' αυτό διστέψαμε την προσέγγιση. Και προτεραιότητα είναι η κατανομή του κέρδους. Εκεί χρειάζονται αλλαγές και ανάλογα με τι αλλαγέ που θα συμφωνήσουμε εκεί μπορεί να αλλάξουμε τους κανόνες του Νέξους. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Όχι, όχι. Καταναλωτές και λοιπά. Όχι. Η FTD. Ο David Coburn. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Φορσόκας είπε στην αρχή σήμερα πως το πιο προφανές είναι το εξή. Είναι απαρχαιωμένη πια η εταιρική φόρη. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτή τη ψύχωση με το να τα φορολογήσουμε όλα. Οι εταιρείε δημιουργούν θέσεις εργασίας, αγορούν, πουλάνε. Και εσείς κάνετε τώρα τούμπες για να φορολογήσετε τις εταιρείε και δεν θα ήταν καλύτερα να μειώσετε την ε, φορολογία ε, ναι. στα μαγαζιά, στο κέντρο, για να μπορούν να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες πάντα θα βρουν παραθυράκια. Και είναι λογική. Και όποιος έχει κάνει επιχειρήσεις στο παρελθόν, ξέρει τι συμβαίνει. Βέβαια, προφανώς αυτό δεν συμβαίνει στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά μόνο ο, ο πολίτης ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσει και να πληρώσει το πλήρε φορολογικό του βάρο. Εγώ νομίζω ότι η κατάργηση του φόρου εισοδήματο ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Οι εταιρείε δεν πληρώνουν φόρους, μετακυλίουν το φόρο στους ε, πελάτες. Άρα λοιπόν τι νόημα έχει όλο αυτό. Δηλαδή, αν κινείται κάτι το φορολογίες και αν εξακολουθεί να μην πεθαίνει, τότε το ρυθμίζεις και νομοθετικά. Ε, νομίζω ότι εντάξει, φίλτρα, ε, λογοκρισία, φόροι, τι, θα βελτιωθεί η ζωή μας έτσι και νομίζετε πως με το να φορολογήσουμε τις εταιρείε θα γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη, δεν νομίζω. Και για ποιο λόγο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλώνει ακόμα περισσότερο κονδύλια για τους χρεοκράτες, για αυτή την κρεατομηχανή νομοθεσίας που έχετε δημιουργήσει. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που πιστεύετε πως οι μεμονωμένες εταιρείε θα σας ακολουθήσουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανείς στην Κομισιόν που να τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Ακόμα και, ο κοινό άνθρωπος τα καταλαβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε εσείς κάποιους από τους επιχειρηματικούς κλάδους για να απαντήσουν σε αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι η ερώτηση σας έχετε να κάνει περισσότερο με το θέμα του κατά πόσο χρειάζεται εταιρική, εταιρικός φόρος ή όχι και όχι με αυτό που συζητάμε εδώ. το κάνετε έτσι για να το κάνετε. Ξέρετε πως δεν μπορεί να τις σε αυτές τις εταιρείε. Πάντα θα βρίσκουν παραθυράκια. Γιατί χάνετε το χρόνο σας. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση για το κατά πόσο τα σύγχρονα κράτη χρειάζονται φόρους για να διατηρηθούν. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα για το τι γίνεται με την ψηφιακή φορολόγηση και εσεί δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό. SND, Mrs. Regner. Ε, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε όλο το πακέτο και για την συνολική, αν θέλετε, παλέτα αυτών των φόρων, φοροσοδήματος, εισοδήματος, η ψηφιακή φορολόγηση. Είναι ένα σύγχρονος τρόπος να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις ε, της τεχνολογίας, της οικονομίας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που μάθαμε χτες από το ΕΚΟΦΗΝ. Δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά και ίσως λίγο πιο σιγά στο Συμβούλιο το θέμα αυτό. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ακριβώς όπως το έχετε προβλέψει. Ο χρόνος φαίνεται να πιέζει, φαίνεται να μην υπάρχει αρκετός χρόνος. Αλλά ποια είναι τα σχέδια, αν θέλετε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο όλες ε, οι διαφορετικές ρυθμίσεις και νομοθεσίες. Και θα σας φέρω μόνο σαν παράδειγμα μία ή δύο που πώς τις αναφέρατε κι εσείς. Υπάρχουν πολλά παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση. Συγγνώμη. πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να έχουμε το ταχύτερο δυνατό συμφωνία. Και γι' αυτό καταβάλουν προσπάθειες. Και η κοινή γνώμη το κατανόησε. Κατάλαβε ότι είναι κατεπήγον θέμα. Πράγματι, προσωρινά μέτρα υπάρχουν. Παραμένουν. Και πολλά άλλα έχουν δρομολογηθεί. Και όλα αυτά αυξάνουν την πίεση για μια δράση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν συνάδελφός μου θέλει να σχολιάσει κάτι. Για την πρώτη ερώτηση δεν είμαστε σίγουροι αν τι πρέπει να πούμε. Το πλήρως πρόγραμμα. Μιλάμε για ψηφιακό φόρο τώρα. Και ορισμός της ψηφιακής εδραίωσης, της ψηφιακής έδρας, εγκατάστασης. Είναι τμήματα Χρειαζόμαστε πληρέστερη προσέγγιση. Αυτά είναι τμήματα, απλώ τμηματικά μέτρα. Πάντηση. Οι κανόνε για την ψηφιακή παρουσία, παρουσία πρέπει να συμπεριθούν στο CCTB και στο CCTB νομικά δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συζητείται στο Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το CCTB ή το CCTB οι προτάσει δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν στο Συμβούλιο και θα ενθαρρύνουμε να εφητηθούν οι κατάλληλοι κανόνες για τη φυσική παρουσία και για την κατανομή των κερδών. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο Catch the Eye, παρόλο που δεν απομένει πολύς χρόνος. Η κυρία Μπερές και η κυρία Γκόμες έχουν ζητήσει το λόγο. Μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα. Η κυρία Μπερές έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στους διερμηνείς που θα μείνω λίγο παραπάνω και μας επιτρέπουν να εκφραστούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να περιμένει στις 10 παρατέταρτο να του δώσουν το λόγο ή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο που να μπορεί να τον πάρει νωρίτερα. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον ΩΣΑ. Μιλήσατε για μια αισιοδοξία η οποία φαίνεται να επικρατεί όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών σας. Δεν πρέπει όμως να να γνωρίσετε ότι υπάρχει μια όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η δράση της Επιτροπής ε, ενισχύει αυτή την αισιοδοξία. Δεύτερον, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας, η έλλειψη πρωτοβουλίας μήπως θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδυαστεί η δική σας δράση με αυτή της Επιτροπής, αντί να προσπαθήσετε να σαμποτάρετε τη δράση της Επιτροπής, να χρησιμοποιήσετε σαν βάση την μέχρι τώρα δραστηριότητα και τις εργασίες της Επιτροπής, έτσι ώστε ο οργανισμός σας να επεξεργαστεί και να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες. Είπατε κύριε Σόργας πως για να αποφύγετε τη διπλή φορολόγηση θα μπορούσατε να σκεφτείτε ένα είδος έκπτωσης ε, ή μείωση στον εταιρικό φόρο. Αλλά αυτό δεν θα έρθει σε αντίφαση με το στόχο της ε, ψηφιακής φορολογίας, για παράδειγμα, με τη ε, την εταιρεία, όπως μια εταιρεία, την Apple, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, που καταβάλει έναν γελίο ε, εταιρικό φόρο και μετά από αυτό θα αφαιρέσετε και το 3%. Δεν μου φαίνεται λογικό. Um, uh, again, we've, first of all, corporate taxes are... Είναι καταρχήν εθνική αρμοδιότητα η φορολογία των επιχειρήσεων και γι' αυτό δεν αποτελεί κομμάτι της προτασής μας. Όμως, αναγνωρίζουμε και ίσως κάποια σενάρια να εμπλέκουν και επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα κράτη-μέλη, άρα λοιπόν που πληρώνουν ε, εταιρικό φόρο στα κράτη-μέλη, που θα πρέπει επίσης να πληρώσουν στο ίδιο κράτος μέλος και το φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γιατί θα εφαρμοστεί σε χώριο επίπεδο λόγω των περιορισμών που έχουμε στις συνθήκες. Δεν υπάρχει πρόβλημα για μας, γιατί ακόμα και οι μη ε, ενωσιακές εταιρείες θα πληρώνουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Δεν πληρώνουν φόρο εταιρικό. Αν δεν πληρώνουν λοιπόν εταιρικό φόρο, από πού θα φερούν το 3%. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχουν φυσική παρουσία ψηφιακή στο κράτος μέλος, δεν φορολογούνται, άρα δεν τους χορηγείται και έκπτωση. επαναλαμβάνω, αν δεν έχει πληρώνει φόρο, δεν θα αφαιρεθεί αυτό το 3%. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη σας ερώτηση. When there is a presence in a member state, um, Όταν είναι παρούσα η εταιρεία, ναι. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ εταιρεών, αν έχουν φυσική παρουσία σε κάποιο κράτος μέλος. Τότε ναι corporate um, um, γιατί ο εταιρικό φόρο που καταβάλλεται δείχνει πως η εταιρεία καταβάλει φόρο στην δικαιοδοσία στην οποία γεννάται το έσοδο. Δεν είναι αυτό το σενάριο που προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε. Λέμε λοιπόν, μια εταιρεία, αν είναι υποκείμενη στους κανόνες για την εταιρικό φόρο, η υπερφορολόγηση με την προσθήκη της, ε, ε, του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει τρέβλωση. Και γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε περιπτώσεις των εταιριών που σέβονται τους κανόνες στη δικαιοδοσία όπου δημιουργείται ε, το έσοδο, μια και οι γενικές, ε, οι γενικοί κανόνες λέει πως φορολογείται το έσοδο εκεί που γεννάται και τη διάκριση με τις άλλες που επιχειρήσεις που ε, δεν είναι φυσικά ε, παρούσες στη συγκεκριτική δικαιοδοσία και δεν υπόκειται σε κανένα είδο φόρο. Όσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις εργασίες μα. Ε, si... Εκ των προτέρων ζητήσω συγγνώμη. Αν αυτά που είπα προηγουμένω, άφησαν να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασιστικό ρόλο συμπεριλαμβανομένη και τη θετική δυναμική που έχουμε εντό τη ομάδα εργασία. Διότι σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλα κάτι κράτη-μέλη αυτής ηγήθηκαν στις συζητήσεις και στο άνοιγμα διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας όπως η Γαλλία με την έκθεση Κολάν Κολάν που είναι έκθεση κινητήρια δύναμη για το θέμα αυτό. Η Γαλλία συμπροεδρεύει στην ομάδα εργασίας και έπαιξε ρόλο κλειδί και παίζει ρόλο κλειδί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλος ιδιαίτερο είναι παρατηρητές εντός ομάδα εργασία και ε, έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα εργασία μα. Ενεργό μέλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ομάδα Εργασία. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και θετικό ρόλο παίζει γενικά και έπαιξε από τη γέννηση του WEPS, ε, BEPS. Θετικό ρόλο όσον αφορά το Digital Service Tax. Πρέπει εκεί να διορθώσω αυτά που είπα, αν θε, άφησα να εννοηθεί ότι θεωρούσα ότι ε, τορπιλίζεται υπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πόρο απέχει αυτή η πρόθεση. Η πρόθεσή μας δεν είναι τέτοια. Εξήγησα αυτά που αναφέρω στην προσωρινή έκθεση, ότι δεν υπάρχει συνένεση όσον αφορά τη χρησιμότητα ενός τέτοιου προσωρινού μέτρου. Αλλά ταυτόχρονα έχουν την κυριαρχία του στα κράτη-μέλη και είναι ελεύθερα και όπως αναφέρεται στην προσωρινή έκθεση, ενδιάμεση έκθεση, να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα που να έχουν μια ισορροπία υπέρ και κατά. Να σταθμίσουν τη χρησιμότητα ενό ε, μέτρου και ενδεχόμενε μελέτε για στρέβλωση ανταγωνισμού προκαλεί κάποιο μέτρο και έτσι να διαφωτίζει το νομοθέτη η σκοπιμότητα ενό μέτρου. Αλλά ουδέμια απόφαση περισκοπιμότητας δεν έχει ληφθεί για ένα τέτοιο μέτρο και όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, ψηφιακό, για το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα συναγάγω συμπεράσματα. Να πω ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση στην Επιτροπή μας το θέμα, στην ΕΚΟΝ. Διαδικαστικός πώς δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες στην Επιτροπή όσον αφορά την σειρά των ομιλητών. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον θέμα σε δημόσια κρόση σε κάποια επιτροπή, πάντα παλεύουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές και να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνειδητή της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τον κύριο Φωσλόγκας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Βανρέη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ρομπέρα από τον ΟΣΑ. Ευχαριστώ τα μέλη, τους διερμηνείς και ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.